Gentlemen, please take your seat. Καθίστε. Welcome our chief election observation. Observe. Καλώς ήρθε και ο επικεφαλής παρατηρητής της αποστολής των εκλογών, ο Γιολάινεν. Πάντα είναι επικεφαλής πάντα είναι επικεφαλής σε χώρες, βασίλεια. Εγώ συνάντησα στη Βεσφαλία το Σάββατο το βασιλικό ζεύγος που ε, ε έλαβαν το βραβείο της Βεσφαλίας ο, ο βασιλιάς Αμπτουλά στο Μούνστερ και το έλαβε μετά Αυτό ήταν ε, βραβείο μετά τη λήξη του πολέμου το 1648 στην, στην Ευρώπη τη ειρήνη της ε, Βεσφαλία. και απονέμεται ε, σε περιπτώσεις πάυσης πολέμου. Εκείνη την εποχή υπήρχε μεταξύ Παρισιού, Βιέννης και Στοκχόλμης πόλεμος μεταξύ αντιπροσώπων όπως τώρα μεταξύ Ριάντ, Τεχεράνης και ίσως και της Άγκυρας. Από τότε δεν άλλαξαν πολλά. Και ίσως ε, αυτή η ειρήνη της, της Βεσφαλίας του 1648 θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδέα για τις χώρες αυτής της περιοχής. Τι σημαίνει να μην ε, υπάρχει ειρήνευση. Η Γερμανία έχασε περίπου το μισό της πληθυσμού μετά από τα 30 χρόνια πολέμου. Είχε λιγότερο από το μισό της πληθυσμό η Γερμανία σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα. Αν δούμε την Μοσούλη, το Χαλέπι, είναι ε, τα ίδια αποτελέσματα του πολέμου. Η αντιπροσωπεία αυτή λοιπόν οι συνάδελφοι Πόχορ Μπέλντα, Ματίας και Δελούντε. Πήγαν να παρακολουθήσουν τις εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες έδρες διατηρήθηκαν από τους μοναρχικούς η αδελφότητα των μουσουλμάνων έλαβε συνολικά νομίζω 60 έδρες. 16 έδρες, συγγνώμη. Ε, μπήκαν στη Βουλή περισσότερα κόμματα, θα μας πει και ο Γιώ Λάινεν και η ε, Μαρία Γκαμπριέλ που ήταν στην αντιπροσωπεία. Ο Γιώ, ευχαριστώ Έλμαρ Χάρηκα που έλαβαν το βραβείο της ειρήνης οι βασιλείς, γιατί ο βασιλιάς είναι εκείνο που προωθεί τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες στην Ιορδανία. Μια χώρα σε μια περιοχή με πολλές συγκρούσεις και ταραχές. Και η Ιορδανία, αν θέλετε, είναι ένα, μια νησίδα σταθερότητας και ειρήνης. Οι βουλευτικές εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν κομμάτι μιας συνεχιζόμενης μεταρρυθμιστικής διαδικασίας που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Και ήταν πολύ σωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε αντιπροσωπεία παρακολούθησης των εκλογών και είμαστε και μια εξαιρετική ομάδα από την και από, την, ε, το Κοινοβούλιο και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρα, ε, πήγαμε από την πρώτη μέρα της προεκλογικής εκστρατείας μέχρι το κλείσιμο της ε, εκλογικής διαδικασίας και εκπονήσαμε τελική έκθεση. Η εκλογές αυτές ε, για το 18ο ε, Κοινοβούλιο συνδυάστηκε με διαδικασία μεταρρυθμίσεων ε, στην νομοθεσία. Νέος εκλογικός νόμος ίσχυσε τώρα στην Ιορδανία και υπήρξε και πράξη για τα πολιτικά κόμματα. Σε προηγούμενες βουλευτικές εκλογές ψήφιζαν προσωπικά προσωπικότητες. Τώρα ε, καταρτίστηκαν εκλογικοί κατάλογοι, ε, ε, μπορεί κανείς λοιπόν να ψηφίσει με βάση το το, κομματικό ψηφοδέλτιο και έχει και μια ψηφοπροτίμηση. Εγώ είχα πάει στη Γκαμπούρ με τη Μαρία Γκαμπριέλ πριν από λίγες εβδομάδες και είχαμε διαφορετικές ε, ε, ιδιότητες, εκείνη ήταν επικεφαλής και εγώ ήμουν εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου. Ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσαν οι αλλαγές να ισχύσουν, καταρτίστηκαν οι κατάλογοι με τους υποψηφίους έγκαιρα και η οργάνωση των εκλογών ήταν καλή. Η προεκλογική εκστρατεία ήταν ήρεμοι, υπήρξαν ε, μικρό ε, παραβιάσεις ε, της διαδικασίας. Κάποια πράγματα δεν έτυχαν του κατάλληλου σεβασμού, αλλά δεν επηρέασαν την έκβαση των εκλογών. Η εκλογική εκστρατεία στην Ιορδανία είναι διαφορετική από αυτά που ξέρουμε εμείς ε, οι εκεί οι υποψήφοι ε, καλούν σε τέντες, σε σκηνές ε, τον κόσμο και προσπαθούν να τους ποιήσουν, να τους ψηφίσουν. Γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. αυτή τη φορά είχαμε ένα σύστημα παθητικής ψήφου. Κάθε πολίτης είχε δικαίωμα ψήφου. Αυτό ήταν διαφορετικό από την προηγούμενη φορά όπου ήταν σύστημα ενεργηγού ψήφου. Έπρεπε κανείς να πάει και να εγγραφεί. Με την αλλαγή του συστήματος αυξήθηκαν κατά 80% οι ψηφοφόροι και αυτό επηρέασε τη συνολική έκβαση. 36% του πληθυσμού ε, προσήλθε στις κάλπες. 200.000 παραπάνω ήταν οι ψηφοφόροι σε σχέση με το 2013. Οπότε μπορεί κανείς να κρίνει ε, ε, αν ήταν επιτυχία. Ήταν επιτυχία αφού αυξήθηκαν κατά 200.000, αλλά το 36% του πληθυσμού σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο κενό, ε, υπάρχει χάσμα μεταξύ συστήματος και πολιτών. Και ήταν λυπηρό το γεγονός ότι οι νέοι απέσχον η Ιορδανία έχει πολύ νέο πληθυσμό, έχω τα στοιχεία, περίπου το 70% είναι κάτω των 30 ετών στην Ιορδανία. Οι νέοι όμως δεν πήγαν στις κάλπες γιατί δυσπιστούν απέναντι στους υποψήφιους και αν αυτοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους και αν είναι σωστό κοινοβούλιο ε, ή αν ε, επιδιώκει άλλα συμφέροντα. Το καλό ήταν ότι δεν μποϊκοτάρισε τις εκλογές κανένα κόμμα. Έχουμε 50 εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα, 39 αμφισβήτησαν τις εκλογές. Όχι, συμμετείχαν σε εκλογές, αλλά οι υπόλοιποι δεν είχαν ε, υποψηφίου, αλλά υποστήριξαν τις εκλογές, οπότε ήταν ειρηνικό το κλίμα, γιατί ε, το Ισλαμικό κόμμα δεν ε, συμμετείχε, αλλά δεν τον μποϊκοτάρισε όπως το 2013. Δεν μποϊκοτάρισε τις εκλογές. Αναφέρατε κι εσείς, κυρία Πρόεδρε, ότι είχαμε μεγάλη συμμετοχή γυναικών στην προεκλογική εκστρατεία και, ε, και στα ψηφοδέλτια και όπως ξέρετε υπάρχουν έδρες ε, ειδικά ε, για γυναίκες και μειονότητες, 15 η κάθε κατηγορία και 5 γυναίκες από τη τώρα είναι 20 συνολικά γυναίκες σε ένα κοινοβούλιο 130 εδρών. Δεν είναι ακόμα μη μεγάλο το ποσοστό, είναι πολύ χαμηλό, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και μάλιστα η ένταξη των νέων ανθρώπων η, θα αυξη, και η αύξηση της ε, συμμετοχής των γυναικών μπορεί να είναι ένας στόχος για το μέλλον. Πολλές οργανώσεις παρακολούθησαν τις εκλογές, ε, η δικά μας η ομάδα ήταν πολύ καλή, καλά προετοιμασμένη, ε, με επαγγελματισμό και υπήρχαν και 30.000 ε, εθνικοί παρατηρητές. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα δηλαδή εθνικό για την παρακολούθηση των εκλογών. διάφοροι έκαναν καταγγελίες, κάποιοι προσέφυγαν και στα δικαστήρια και είδαμε ότι τα δικαστήρια ήταν αμερόληπτα και έγκαιρα εξέδιδαν τις αποφάσεις τους. Θα έλεγα ότι αυτές οι εκλογές στην Ιορδανία συνιστούν περαιτέρω βήμα ανοίγματο της χώρας, στις ε, διαδικασίες των μεταρρυθμίσεων. Βέβαια, Είδαμε κάποιες ιδιαιτερότητες που αναφέρομαι στις συστάσεις. Τα μέσα ενημέρωσης δεν εκάλυψαν την προεκλογική εκστρατεία, δηλαδή ενημέρωσαν ότι διεξάγονται εκλογές, αλλά δεν ενεπλάκησαν στην προεκλογική εκστρατεία. Και θεωρήσαμε ότι είναι μερική μόνο η ελευθερία τον ΜΜΕ. Μήπως υπάρχει αυτολογοκρισία, σκεφτήκαμε. Φοβόντουσαν πως κάνουν κάτι λάθος, οπότε δεν κάλυψαν τις συνεδριάσει ε, και τις εκδηλώσεις και αυτό είναι ένα έλλειμμα. Υπήρχαν επίσης περιοχές ε, αγροτικές που υπερεκπροσωπούνται ενώ αστικές περιοχές υποεκπροσωπούνται και η κατανομή των εδρών δεν ε, ε, συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και η ισότητα ε, ψήφου δεν είναι εγγυημένη. Στο Αμάν, ας πούμε, οι έδρες είναι λιγότερες στην περιοχή εκείνη από τις ισχυωρικές περιοχές, τις αγροτικές. Και για να είναι κανείς υποψήφιος υπάρχουν κάποιες περιοριστικές διαδικασίες εγγραφής, πρέπει κανείς να καταβάλει κάποια χρήματα και στο τέλος οι περισσότεροι υποψήφοι είναι από φυλές, επιχειρήσεις ή πρώην βουλευτές. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος λοιπόν γιατί οι νέοι έχουν κάποιες επιφυλάξεις ε, απέναντι σε αυτές τις εκλογές και δεν συμμετέχουν. Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι η αρχή για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Εμείς τις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλουμε την επίσημη έκθεση, αλλά αυτά ε, προς το παρόν για την ενημέρωση των μελών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζουλένιν και την ομάδα του για την εξαιρετική δουλειά τους. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε και την υποδοχή και επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χάρη στο δουλειά των οποίων μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώ αυτή την αποστολή. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα θετικά σημεία γιατί θα πρέπει να τα τονίσουμε. Είχαμε μια καταρχήν θετική εμπειρία και όπως είπε και ο επικεφαλής, καταρχήν ήταν η διαδικασία διαφανής και ε, του συμπεριλαμβάνε όλους και ε, την ε, ημέρα των εκλογών ε, διεξήχθησαν εκλογέ με ρομοτρόπο. Υπήρχαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά βέβαια, αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Έχουμε δύο σημαντικού παράγοντε. Δηλαδή, έχουμε αφενό στο πλαίσιο μια φιλόδοξη πολιτική μεταρρυθμίση και από την άλλη έχουμε μια ασταθή περιφερειακή κατάσταση όπου υπάρχουν απειλές ασφαλείας. Τώρα θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία κλειδιά. Καταρχήν, είχαμε μία αποστολή η οποία βασίζεται στο έργο της αποστολής που έστειλε η Ένωση το 2013. Ακολουθήθηκαν οι συστάσεις. Αυτό πρέπει πάντα να το λέμε, γιατί δεν ισχύει σε όλες τις χώρες όπου μεταβαίνουμε. Κατόπιν είχαμε τις πρώτες εκλογές με νέο εκλογικό νόμο, που στοχεύουν να ε, βοηθήσουν την ανάδεση ενός πολυκομματικού συστήματος. Ε, βέβαια είδαμε ότι η ψηφοφορία συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να καθορίζεται από τη φυλή, τη θρησκεία στην οποία ανήκει ο καθένας. Έτσι λοιπόν είχαμε πρώτη φορά πραγματικά πολιτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν από τα κόμματα ε, και φυσικά και στα πλαίσια της Νέας Συνέλευσης και εμεί έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε συζητήσουμε στη συνέχεια. Υπόθηκε επίσης, ε, είχαμε το νέο κατακαιρματισμό και το διαχωρισμό των εκλογικών περιφερειών. Κάποιες ε, αστικές περιοχές ε, είναι υποεκπροσωπούμενες, ενώ κάποιες περιοχές της επαρκείας υπερεκπροσωπούνται. Και θα ήθελα τώρα να επιμείνω στην εκλογική αποστολή και θα ήθελα να αναφέρω στην εξάρτητη εκλογική επιτροπή ήταν καλά οργανωμένη και διαφανής. Βέβαια δεν δημοσίευσε τις αποφάσεις της ε, για τις έγκυρες υποψηφιότητες ή τις μη έγκυρες ε, και σε περίπτωση που απορρίπτεται κάποια ψηφιότητα δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν ένδικα μέσα σε δεύτερο βαθμό. Επίσης ε, ήταν το σύστημα ψηφιοποιημένο, αυτό ήταν κάτι πολύ θετικό και έδωσε ε, ουσιαστικά θετική εικόνα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία συζήτηση στην οποία μπορούν να συσφέρουν τα μέσα ενημέρωσης για να μπορέσουν να επιλέξουν οι πολίτες σε βάση των ιδεών και των σχεδίων των κοινωνικών που παρουσιάζονται. Και θέλω να επιμείνω σε δύο μεγάλε κατηγορίε ε, τη κοινωνία, του νέου και τι γυναίκε. Καταρχήν, για τι γυναίκε μεγάλη δουλειά πρέπει να γίνει, γιατί παρά το σημαντικό αριθμό των γυναικών που συμμετείχαν, εξακολουθούν να πρέπει να γίνει δουλειά και από τα μέσα ενημέρωση ε, σε, ό,τι αφορά ε, την διαφοροποίηση μεταξύ του θέματος γυναίκες ποσοστός και γυναίκες υποψήφοι. Επίσης, ε, για τους νέους πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να κινητοποιηθούν, να μπορούν ε, να έχουν κάποια κίνητρα να πάνε στις κάλπες και φυσικά από την πλευρά τους πρέπει να το γνωρίσουμε ότι όταν εμείς πήγαμε στα εκλογικά κέντρα είδαμε ότι σχεδόν κανένας νέος δεν υπήρχε εκεί να ψηφίσει και είδαμε ότι ούτε ε, και οι ντόπιοι βοηθοί μας ήθελαν να ψηφίσουν. Δηλαδή παραμένουν επικριτικοί και πρέπει να δουν ποια κατεύθυνση θέλουν να δώσουν στην ανάπτυξη της χώρας τους. Αυτά ήταν τα κυρία σημεία που θέλω να αναφέρω εγώ και συμπερασματικά να επιμείνω στο εξή. Εμείς ω Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και πολιτικά και τεχνικά αυτές τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του εκλογικού κύκλου και πέραν αυτού. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για να γίνει η δημοκρατική μετάβαση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τέθηκαν οι βάσεις και χάρη σε αυτές τις εκλογές και μέσα τη συνεργασίας θα προχωρήσουν τα πράγματα και γενικά υπήρχε μια συνολική θετική εικόνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Πρέντα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας για την παρουσίαση που μας κάνανε, τις αποστολής παρακολούθησης των εκλογών στην Ιορδανία. Δύο ερωτήματα έχω. Το πρώτο αφορά την συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές. Θυμάμαι ότι στις προηγούμενες εκλογές, όταν ήμουν και εγώ παρατηρητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι γυναίκες είχαν προσκληθεί να ψηφίσουν σε χωριστά εκλογικά τμήματα και από ό,τι θυμάμαι είχε υπάρξει μια πολύ καλή συμμετοχή γυναικών στις εκλογές. και πάλι και στις τρέχουσες εκλογές ήταν μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών από τη συμμετοχή των ανδρών. Ο Γιώ Λάινεν ανέφερε ότι δεν έγινε από την ε, μια <clears throat> πληροφοριακή εκστρατεία για τις εκλογές. Δεν ξέρω αν δόθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί προς τον πληθυσμό. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που ήταν ε, κύριος παρατηρητής ο Ντέβιτ Μάρτιν, ότι είχαμε εκπλαγεί γιατί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ήρθαν στη συνέντευξη τύπου δεν έθεσαν κανένα ερώτημα. Η μόνη συνέντευξη τύπου που έχω ζήσει όπου κανείς δεν ρώτησε τίποτα. Ε, έγινε απλώς μια παρουσίαση χωρίς ε, αντίδραση από τους ε, δημοσιογράφους. Δεν ξέρω αν, έχουν απλώς, αν κατέγραψαν απλώς τα σχόλια μας οι δημοσιογράφοι αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή τη φορά υπήρξαν δημοσιογράφοι που να θέσουν ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι αν υπάρχει πραγματικά μια πληροφόρηση προ τον πληθυσμό ότι έχουμε αυτά τα κόμματα, τότε θα γίνουν οι εκλογές, αυτή είναι η υποψήφη κτλ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Όταν είχαμε πάει πριν από ένα μισό χρόνο στο Μεξικό, δεν υπήρξαν και εκεί ε, ε, ερωτήσεις από τους ε, δημοσιογράφους. Και αυτοί οι οποίοι ρωτούσαν ήταν άτομα τα οποία ήταν υπάλληλοι του Κοινοβουλίου, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είχαν προσκαλέσει δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου. Αυτό ήταν μία από τις κορυφώσεις της πολιτικής μου καριέρας, κατά κάποιο τρόπο. Θέλει κάποιος άλλος να, να λάβει το λόγο. Όχι. Ευχαριστώ. το θεσμικό <clears throat> κόμμα της Επανάστασης είναι αυτό που είχε την εξουσία τότε στο Μεξικό. Ωραία. Κάνουμε λοιπόν μια σύντομη διακοπή. Α, μια στιγμή ο γιο. Ναι, ε, αγαπητέ συνάδελφε Πρέντα, όταν ξεκίνησε η αποστολή εκλογικής ε, παρακολούθησης ήταν ακριβώς όπως το είπατε, δεν ρώτησαν καθόλου όταν είναι παρουσία πριν από την, ε, τις εκλογές δεν είπαν τίποτα οι δημοσιογράφοι. Μετά από τις εκλογές ήταν πιο πολλοί δημοσιογράφοι από ξένα μέσα ενημέρωσης από ότι εθνικοί δημοσιογράφοι. Λίγα πράγματα ρωτήσαν, όχι πολλά. Υπάρχει μια αυτολογοκρισία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία του, των μέσων ενημέρωσης είναι κάτι το κάπως περιορισμένο στην Ιορδανία. Ναι, οι γυναίκες <clears throat> πράγματι ψηφίζουν χωριστά από τους άνδρες. μόνο τούτο, από τα 1,5 εκατομμύρια ψηφοφόρων που ήρθαν στις εκλογές, ήταν 58% ε, οι γυναίκες και 42% οι άνδρες. Ψήφισαν λοιπόν χωριστά οι γυναίκες, αλλά ήταν μεγάλη η συμμετοχή τους η Εκλογική Επιτροπή επίση έκανε πολλά πράγματα για να μπορέσει να πληροφορήσει τον πληθυσμό, αλλά τα μέσα ενημέρωση θα μπορούσαν να έχουν δώσει και περισσότερε ειδήσει σε σχέση με την εκλογική διαδικασία. Και εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε η <clears throat> Μαρία Γκάμπριελ λέγοντα ότι όπω είπε σωστά πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθήσει περισσότερο την εκλογική διαδικασία στην Ιορδανία. Είναι μια σημαντική χώρα για την ασφάλεια της περιοχής. Όπως ε, είπα και στο Twitter, η Ορδανία έχει 10 φορές περισσότερους πρόσφυγες ε, κατά κεφαλή από τη Γερμανία και πολύ λιγότερα κονδύλια. Γι' αυτό πήρε και το βραβείο ο βασιλιάς Αμπτουλάχ γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό ε, προσφύγων και πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους για να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν ήταν καθόλου θέμα στην ε, προεκλογική εκστατεία. Ευχαριστώ. Dear colleagues, we will start in a minute the meeting with Devon. Mr. McEwan is approaching and will chair. Κύριε Μακιούαν και θα συμπροεδρεύσει στη συνεδρίαση αυτή.